επαφή με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Λοιπόν, υπάρχει μία πρόταση πέντε ομάδων, παράγραφος 1, αρχικό κείμενο, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3, ε, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα με ονομαστική άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται το κείμενο. Τέταρτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Το κείμενο εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται το κείμενο. Έκτο τμήμα με ονομαστική και πάλι άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται το κείμενο. Μετά την παράγραφο 3, 2 με ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται το κείμενο. Τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 4 τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία με ονομαστική. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Το κείμενο εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Το κείμενο εγκρίνεται. 4. Στην παράγραφο 5 με ονομαστική ψηφοφορία η οποία και αρχίζει. Πέρας. Το κείμενο απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο με ονομαστική η οποία και αρχίζει. Πέρας. Το κείμενο εγκρίνεται. Παράγραφος 6 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα με ονομαστική άρχεται. Πέρας. Το κείμενο εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα άρχεται. Πέρας. Το κείμενο εγκρίνεται. 5 στην παράγραφο 7. Άρχεται η ψηφοφορία με ονομαστική. Πέρας. Το κείμενο απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Το κείμενο εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται το κείμενο. Τρίτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται το κείμενο μετά την παράγραφο 7, τροπολογία 6 με ονομαστική οποία και αρχίζει. Πέρας, το κείμενο απορρίπτεται. Τροπολογία 7 με ονομαστική άρχεται. Πέρας, απορρίπτεται το κείμενο. Παράγραφος 8, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Αρχικό κείμενο σε τέσσερα τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική η οποία και αρχίζει. Πέρας. Το κείμενο εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα με ονομαστική οποία και αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται το κείμενο. Παράγραφος 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 10, τροπολογία 8 με ονομαστική άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται το κείμενο. Τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Το κείμενο απορρίπτεται. Παράγραφος 11. Αρχικό τμήμα. 1. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παραγραφός 12 αρχικό ε, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παραγραφό 12 τροπολογία 10 με ονομαστική η οποία και αρχίζει. Πέρας. Απορρίπτεται το κείμενο. Τροπολογία 11, πάντα με ονομαστική, η οποία και αρχίζει. Πέρας, το κείμενο απορρίπτεται. Παράγραφος 13, αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 14, δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράχρος 15 τροπολογία 12 με ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται το κείμενο. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Ε, παρακαλώ, ονομαστική με συγχωρείτε. Πέρας, εγκρίνεται το κείμενο. Μετά την παράγραφο 15, τροπολογία 13 με ονομαστική, η οποία και αρχίζει. Πέρας, απορρίπτεται α. Άρχεται η ψηφοφορία του αυθεντικού κειμένου, του αρχικού κειμένου. Πέρας. Εγκρίνεται το κείμενο αιτιολογική σκέψη β υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται αιτιολογική σκέψη σ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται Δ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το H, τροπολογία 1, με ονομαστική η οποία και αρχίζει. Πέρας. Το κείμενο απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την πρόταση ψηφίσματος με ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται το κείμενο. Συγχαρητήρια στους συντάκτες. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, επιτρέψατε μου να σας κάνω μια μικρή προσωπική δήλωση. Ορισμένοι από εσά γνωρίζετε ότι είμαι υποψηφία για την ομάδα, των Πρασίνων. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα εγκαταλείψω το Κοινοβούλιο και είναι η τελευταία ε, ψηφοφορία της οποίας ε, προεδρεύω εγώ ως Αντιπρόεδρος και θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω και θα ήθελα να πω ένα μικρό ευχαριστώ για αυτά τα 8 χρόνια που συνεργάστηκα με πολλούς από εσά σε αυτό το κοινοβούλιο ε, συμμεριζόμενοι το πνεύμα της ε, συνεργασίας το οποίο καλλιεργούν τουλάχιστον περισσότεροι από εσά σε αυτό το σώμα και επίση αυτά τα τρία χρόνια ω μία των αντιπροέδρων. Ήταν πολύ γόνιμα αυτά τα χρόνια για μένα και σα υπόσχομαι ότι πραγματικά θα κομίσω αυτό το ευρωπαϊκό πνεύμα το οποίο βίασα εδώ στις, στο εθνικό επίπεδο και στο Αυστρικό Κοινοβούλιο και πραγματικά αναμένω με ανυπομονησία τη μελλοντική μα συνεργασία υπό μια διαφορετική μου ιδιότητα γιατί χρειαζόμαστε ισχυρά εθνικά κοινοβούλια και ένα ισχυρό ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Σε ευχαριστώ πολύ και τώρα θα περάσουμε στις ψηφοφορίες. Η πρώτη είναι η έκθεση της κυρίας ε, Βαλεάν, ο περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό, ε, τροπολογία υπαριθμών 5, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου έχει ολοκληρωθεί. Και τώρα περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία για την έκθεση του κυρίου Μάτο όσον αφορά τα μέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζει στη ζώνη της Σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη διατήρηση των θηνοειδών. 34 ε, άρχεται η ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Και τώρα θα περάσουμε στην τροπολογία υπαρχών 33, αντιδρατάσεις των χειρών, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και εδώ ολοκληρώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Η επόμενη ψηφοφορία είναι η έκθεση της κυρίας ΣΑΕΤ για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράγραφος 2 του αρχικού κειμένου, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 9 του αρχικού κειμένου, διανατάσεις των χειρών, υπέρ, κατά, αποχές, επίσης εγκρίνεται. Παράγραφος 15 του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα, το πρώτο τμήμα με ανομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η δεύτερη παράγραφος, επίσης με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Ρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 19 του αρχικού κειμένου, ε, ψώνοντας το χέρι, υπέρ, κατά, αποχές, Ηλεκτρονική επαλήθευση, παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 21 του αρχικού κειμένου, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 23 του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Παράγραφος 25 του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα. Το πρώτο υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Παράγραφος 27 του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές θα λέγω ότι εγκρίνεται παράγραφος 28 του αρχικού κειμένου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 31 του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές επίσης εγκρίνεται. Παράγραφος 35 του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα με ονομαστική ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 39 του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, θα ήθελα να γίνει επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 42 του αρχικού κειμένου υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 44 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 45 του αρχικού κειμένου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 48 σε δύο τμήματα του αρχικού κειμένου το πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 52 του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος, ας γίνει θευσή. Παράγραφος 52, δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 56 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Συγγνώμη. Με συγχωρείτε. Ε, παράγραφος 55 του αρχικού κειμένου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαλήθευση. Καλώς. Παράγραφος 55 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Παράγραφος 56 με ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 57 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα, για τάσσουν στο χειρόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ωραία, επαλήθευση, αλλά νομίζω ήταν ξεκάθαρο. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας, απορρίπτεται. 59 το αρχικό κειμένο υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Παράγραφο 61 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα με νομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 62 μονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 63 το αρχικού κειμένου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη. Δέλτα. Ε, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εταλογική σκέψη S σε δύο τμήματα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, επίσης εγκρίνεται. Ε, σκέψη AD. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και τώρα θα έρθουμε στο ψήφισμα στο σύνολό του με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στους συγγητές. Ε, στον εισηγητή, συγγνώμη. Επόμενη έκθεση είναι της κυρίας Τερέζα Μπάριο, διαδικαστικό. Please try again, try again. Ε, αν μπορείτε, παρακαλώ, ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Ναι. Στο συγγνώμη, κύριε συνάδελφοι, αλλά δεν παίρνω συχνά το λόγο για κάτι διαδικαστικό. Όμως, χρειάζεται. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το σύστημα ψηφοφορία τη θέση μα εδώ πάνω. Μήπω μπορεί κάποιο τεχνικό να το ελέγξει, παρακαλώ. Η πρόεδρο, θέλετε να έρθει κάποιο από την τεχνική υπηρεσία. Ναι, θα παρακαλέσω, αν μπορεί, ε, να ελέγξει το σύστημα ψηφοφορία στη θέση του κ. Κάλβα. Ωραία. Α προχωρήσουμε τώρα στην ψηφοφορία για την έκθεση τη κυρία Τέρα Αχημένε Δερφίλ Μπάριο, αντιμετώπιση τη συρρήκνωση του χώρου τη κοινωνία των πολιτών στι αναπτυσσόμενε χώρε. Ξεκινώντα από την παράγραφο 5, με ανάταση το υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Δεύτερο μέρο, υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται επίση. Α ελέγξουμε ηλεκτρονικά Θέλετε δεύτερο μέρος λοιπόν της παραγράφου 5. εν, άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. ψηφοφορία. Όχι. Εγκρίνεται. 9. Με ανάταση χειρός, αρχικό κείμενο υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 σε δύο μέρη. Για το πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο μέρο υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται επίση. 23, αρχικό κείμενο, υπέρ, κατά, Αποχέ. Α ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ, για την παραγραφή 23, ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Με μικρή διαφορά, αλλά απορρίπτεται. 32 για το πρώτο σκέλος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Για το δεύτερο σκέλος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται επίσης. Παράγραφος 36, αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Για το ψήφισμα, συνολικά, με ε, ονομαστική κλίση και ηλεκτρονικά ψηφίστε παρακαλώ. The vote is closed και εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Επόμενη ψηφοφορία. Έκθεση της κυρίας Βόζενμπεργκ Βριονίδη κατά πολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων. Παραγράφος 38, αρχικό κείμενο, με ανατεσχυρός υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 78 αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη π. Αρχικό κείμενο. Θέλετε να ελέγξουμε για την 78 ηλεκτρονικά βεβαίως. Ε, παράγραφος 78 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται αιτιολογική σκέψη π, αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Με παρόμοια πλειοψηφία, αλλά σε ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Αιτιολογική σκέψη π, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Για το ψήφισμα συνολικά με ονοματιστική κλίση ψηφίστε παρακαλώ. The vote is... Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. The Επόμενη ψηφοφορία από τον κύριο Μπιουτικόφερ. Πολιτικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον ΑΖΕΑΝ. Ε, υπάρχει μία τροπολογία ή ένα από τον εισηγητή με ανάταση χειρός υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και για το ψήφισμα στο σύνολό του με ονομαστική κλίση. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. The vote Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια για τον εισηγητή. Ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και καλή όρεξη σε όσους αποχωρήσουν. Dear Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους που αποχωρούν από την αίθουσα να το κάνουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία επεξήγησης ψήφου. dear colleagues we will start with the explanation of votes and the από τη συνάδελφη θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία τη λόγηση ψήφου, ξεκινώντα από του ομιλητέ που έχουν ζητήσει το λόγο για την, το ψήφισμα για την πορεία διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο.